Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 135 του κανονισμού. Λάμπερτ. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Τα συλληπιτήριά μας, εγώ και των συναδέλφων μου, στους φίλους και συγγενείς αυτών που έχασαν τη ζωή τους στη Λαχώρη στην εορτή του Πάσχα. Τα συλληπιτήριά μας επίσης και στα θύματα όλων των άλλων επιθέσεων στη χώρα αυτή. Υπάρχει μια αύξηση των επιθέσεων από πλευράς των ε, ακεραιοφρόνων με δύο τρόπο Βέβαια είναι θετικό το μέτρο της κυβέρνησης ε, να βελτιώσει την διδακτέα ύλη των σχολείων με περισσότερη επιμονή στον σεβασμό των θρησκευτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαιτεί και τη δημιουργία μιας πλήρως ανεξάρτητης Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. και στα πλαίσια της Συμφωνίας ε, και Πασίν. Επίσης θα πρέπει να επανεξεταστεί και ε, το θέμα της κατάργησης της θανατικής ποινής. Βίντεν Χόλτζερ είναι στην αίθουσα. Όχι, τότε περνάμε στον κύριο Κέλαμ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ανησυχούμε για την ε, συνεχιζόμενη βία στο Πακιστάν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εταίρο Ευρωπαϊκής Ένωσης Στη Λαχώρη 24 Μαρτίου η επίθεση κατά των χριστιανών. Στα τα περισσότερα δήματα ήταν μουσουλμάνοι και εκφράζουμε τη λύπη μας προ όλα τα θύματα. Όμως δεν είναι εξαίρεση η Λαχώρη. Υπάρχουν συστηματικέ παραβιάσει ε, τη ε, ανεξιθρησκείας για, όλες, για όλου του χριστιανού, Σουνίτε ή ειδουιστέ και πλήτουνται οι μειωνότητε από διακριτική μεταχείρηση θεσμοθετημένοι μέσω τη νομοθεσία. Υπάρχουν όμω περιβλασφημία που πλείται ιδιαίτερα αυτή τη μειωνότητε, Σουνίτες, Ινδουιστές και πλήττονται οι μειονότητες από διακριτική μεταχείριση με θεσμοθετημένη μέσω της νομοθεσίας. Ε, ε, υπάρχει ο νόμος περί βλασφημία που πλήττει ιδιαίτερως αυτές τις μειονότητες. Η Άση Σαμπίμπη η οποία κατηγορήθηκε, καταδικάστηκε σε θάνατο λόγω βλασφημίας και έξι χρόνια τώρα κρατείται. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ζητήσουμε άμεση απόδοση της δικαιοσύνης στην περίπτωσή της και είναι κοινή μας ανησυχία η τύχη των θρησκευτικών μειονοτήτων και ζητούμε από την ύπατη εκπρόσωπο Μογκερίνη να συνεργαστεί με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν για την καταπολέμηση της μυσαλλοδοξίας και της τρομοκρατίας. Ο κύριος Uh, για όσους ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες ε, στο Πακιστάν η ζωή μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους ε, Αμεντίς, ε, τους Ινδουιστές, τους Σιήτες και κυρίως για τους Χριστιανούς. Η αποτρόπια τρομοκρατική επίθεση της Ελλαχώρης δυστυχώς δεν είναι μονομένο συμβάν και θα πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα από το Κοινοβούλιο. Θα ήταν άδικο να πούμε ότι δεν έχει αναλυθεί καμία δράση. Παρόλα αυτά ζητώ από την πακιστανική κυβέρνηση να κάνει περισσότερο τόσο ώστε να επικρατήσει η ανεξιθρησκεία και ανεκτικότητα προ όλε τι θρησκευτικέ μειονότητε. Υπάρχει αδυναμία για να αντιμετωπιστεί αυτή η νομοθεσία για τη θρησκεία. Ε, Νόμο βλασφημία, παραδείγματο χάρη, σχετικά διατάγματα θα πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία ε, κατά προτεραιότητα. Ο Άσυση που ζήτησε καταργησή της, ε, του νόμου περί βλασφημίας και το πλήρωσε με τη ζωή του θεωρείται ήρωα από πολλού πακιστανού. Ε, και ε, υπάρχουν ε, εξτρεμιστικά ρεύματα στο Πακιστάν. Δυστυχώ αυτό διαπιστώνουμε. Η μυσαλλοδοξία έχει διαπιστωθεί σε πάρα πολλέ περιπτώσεις και ελπίζω να υπάρξει βούληση για αλλαγή στην κυβέρνηση και στο λαό του Πακιστάν. Ευχαριστούμε κύριο Βάτσινχολτσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το Πακιστάν στα κατεπήγοντα. Και πάντα το θέμα είναι η θρησκευτική... τα θρησκευτικά προβλήματα. Βεβαίω οι Ταλιμπάν είναι μια τρελή σέχτα που έχουν μια δική του ερμηνεία του Ισλάμ και βεβαίως ε, οι πιο ήπιοι μουσουλμάνοι αλλά και οι άλλες θρησκείες είναι ο στόχος τους. Αυτή τη φορά ο στόχος ήταν οι χριστιανοί, ε, θύματα ήταν και άλλοι μουσουλμάνοι. Πρόκειται για κάτι το αποτρόπαιο και εγκληματικό. Και θεωρώ πως πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αδρανοποιηθεί αυτή η απειλή και να αναμένουμε το Πακιστάν να κινητοποιηθεί ε, σοβαρά κατά αυτής της απειλής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βερζιά έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η απόπειρα στο Λούνα Πάρκ της Λαχώρης προκάλεσε πάρα πολλά θύματα. Οι ένοχοι είχαν σαν στόχο τους χριστιανούς, αλλά η πλειοψηφία των θυμάτων ήταν μουσουλμάνοι. 15 μέρες πριν είχαν χτυπήσει τα σιητικά τεμένη. Υπάρχουν εντάσεις στο Πακιστάν και οι ρίζες βρίσκεται και στην πολιτική της πακιστανικής κυβέρνησης η οποία στην αρχή χρηματοδότησε τοποκρατικές ομάδες οι οποίες είναι εκτός ελέγχου πλέον αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες του Περσικού. Τα στρατιωτικά δικαστήρια, ο νόμος περί βλασφημίας, θα πρέπει κανονικά ε, το Πακιστάν στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με την Ένωση να βελτιώσει τις επιδόσεις του. Ξέρουμε τον ιστορικό ρόλο του Πακιστάν στην αποσταθεροποίηση της περιοχής. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πιέσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Τέλος. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η επιθέση στην Λαχώρη ήταν μια αποτρόπια επίθεση στο λαό του Πακιστάν και σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει τα συλληπιτήριά του και την στήριξή του στις οικογένειες των θυμάτων και των τροματιών. Όμως πρόκειται για άλλη μία δυστυχώς ε, επίθεση και δεν υπάρχουν σημεία βελτίωσης. Πρέπει τώρα το Πακιστάν να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και να αντιμετωπίσει τη θρησκευτικό εξτρεμισμό γιατί ξανά, αλλιώς ξανά και ξανά τα ίδια θα λέμε γι' αυτό σήμερα ζητάμε από τις αρχές του Πακιστάν να περάσουν στον ιδεολογικό αγώνα κατά του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας αλλά και να αντιμετωπίσουν και την, ε, τον κοινωνικό αποκλεισμό Ας είμαστε σαφείς. Όμως δεν θα πετύχει μόνο του το Πακιστάν. Χρειάζεται μπλοκή όλων ε, των χωρών της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας. Τέλος, εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε και εμείς ένα ρόλο να παίξουμε. Γι' αυτό ζητάμε σήμερα την κυρία Μογκερίνη και το Συμβουλίο να έρθουν σε επαφή με την κυβέρνηση του Πακιστάν για να αντιμετωπιστεί η απειλή τη τρομοκρατία και να βοηθήσουν τον πακιστανικό λαό στι ε, προσπάθειε του για να εξαλείψει την τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά του εισηγητέ, ε, περνάμε στου ομιλητέ από τι διάφορε ομάδε. Τον λόγο έχει ο κύριο Πρέντα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τρομοκρατική επίθεση στη Λαχώρη στις 27 Μαρτίου, εκείνη τη μέρα όπου οι χριστιανοί όρταζαν το Πάσχα, ε, είναι μια αποτρόπια πράξη Φυσικά ο βασικός στόχος ήταν η χριστιανική κοινότητα, πλην όμως ε, τα θύματα ε, προέρχονται από διάφορες θρησκευτικές ομάδες του Πακιστάν. Ο θρησκευτικός ε, εξτρεμισμός οδηγεί σε τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις και γι' αυτό η καταπολέμηση τρομοκρατίας της πακιστανικής κυβέρνησης θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν άγριο γονά κατά ακριβώς αυτού του φαινομένου του θρησκευτικού εξτρεμισμού. Η πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση αποδεικνύει πόσο απαραίτητο είναι αυτό. Χρειάζεται ανεκτικότητα προς θρησκευτικέ ε, μειονότητες, ε, οι θρησκευτική ανεξιθρησκεία κατοχυρώνεται ε, στο Σύνταγμα όπως και η ελευθερία έκφρασης. Όμως αυτή ο νόμος βλασφημία σε βάση της οποίας καταδικάστηκε η Ασίνα Μπίμπη αναιρεί αυτή την συνταγματική διάταξη. Ευχαριστώ κύριος Χάουιτ. Ε, νιώθουμε το σόκο των τρομοκρατικών επιθώσεων στις Βρυξέλλες και στο Παρίσιας. Ε, θυμόμαστε λοιπόν ότι μόνο το 0,5% των θυμάτων δημοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη ε, και ε, μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια το 20% των δολοφονηθέντων είναι και οι ίδιοι μουσουλμάνοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο στόχος στη Λαχώρη το Πάσχα ήταν ένας παιδικός σταθμός σε μια παιδική χαρά και τελικά επλήγησαν οι πλέον αθώοι. Στις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε κατά της τρομοκρατίας ε, φαίνεται ότι υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ίδια λέμε προς τους φίλους του Πακιστάν μέσα στην, ε, στο ψήφισμα μας. Ζητάμε και πάλι από το Πακιστάν να επανεξετάσει ε, την, ε, τις περιπτώσεις ε, αυτών που έχουν καταδικαστεί βάσει του νόμου της βλασφημίας και ζητούμε την χάρη στην περίπτωση του Ανού Φασέτε και πιστεύουμε ότι όχι μόνο με το Πακιστάν αλλά και σε συνεργασία με όλες τις χώρες που θρηνούν για αυτά τα θύματα θα πρέπει να υποστηρίζουμε τις ίδιες αξίες. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Μπέλτερ. Πρέπει να φύγουν όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στα σχολικά βιβλία του Πακιστάν για τους χριστιανούς και τις άλλες μειονότητες. Και έχουν δίκιο αυτοί που το ζητάνε αυτό, γιατί πρόκειται για δηλητηρίαση του μυαλού της πακιστανικής νεολαίας. Και ερωτώ, δίνουμε λεφτά στο Υπουργείο Παιδείας του Πακιστάν και αν ναι, τι απαιτήσει έχουμε σε αντάλλαγμα. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη παρακολούθηση και των Ισλαμικών ιεροδιδασκαλίων στη χώρα. Προτείνω λοιπόν η Άζια Μπίμπη και οι υπόλοιποι που έχουν κατηγορηθεί για βλασιμία να αφαιθούν ελεύθεροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δέχεστε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Φρουντσουλίκα. Ναι, παρακαλώ. Αγαπητέ συνάδελφε, πέρα από τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις. Ξέρετε πως πολλοί κόσμος φεύγει από το Πακιστάν και έρχεται στην Ευρώπη. Πέρα από τους Σύριους, ε, Αφγανούς και Ιρακίνους. Δεν θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση του Πακιστάν για να σταθεροποιήσει τη χώρα για να μείνει ο κόσμος εκεί. Γιατί ο αριθμός ε, των μεταναστών από το Πακιστάν αυξάνεται καθημερινά. Κύριε Μπέλτερ, συνάδελφε, έχω ασχοληθεί καιρό με το Πακιστάν και λένε ότι υπάρχουν δύο κράτη. Δηλαδή, το, το πολιτικό κράτος και οι στρατιωτικές και θρησκευτικές αρχές. Ε, πραγματικά πρόκειται για μια εκρηκτική κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του γύρου. Λοιπόν, κύριε Χέλβενη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ένα πράγμα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Στο Πακιστάν είχαμε ένα χτύπημα κατά που γιόρταζαν το Πάσχα. Πρέπει να λήξουμε την αλληλεγγύη μας με τα θύματα και τους συγγενείς τους. Εκτελέστηκαν στοχευμένα και οι Ταλιμπάν θέλουν να τους εμποδίσουν από το να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Οι διάφορες ομάδες των Ταλιμπάν ισχυροποιούνται συνεχώς. Η κυβέρνηση προσπαθεί να τους ε, σταματήσει αλλά δεν τα καταφέρνει. <coughs> Υπάρχει όμως ελπίδα. Μετά το χτύπημα ιδρύθηκε το λεγόμενο κίνημα της ανοχής. Το Πακιστάν και η Ευρώπη θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό πιο σοβαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Κάν έχει το λόγο για Πρόεδρε, καταδικάζουμε την επίθεση της Λαχώρης και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες η χώρα αυτή υποφέρει. 60.000 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τέτοιες ενέργειες. 10 δις α, ε, α, ε, ε, λίρες απώλειες στην οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα απαιτείται να υποστηρίξουν την οικονομική αλλά και την πολιτική δράση του Πακιστάν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είδαμε τι συνέβη με την τρομοκρατία στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Δεν είναι σύγκρουση πρόβλημα ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες ή σε διαφορετικές θρησκείες. Απλά οι εξτρεμιστές θέλουν να διαλύσουν το καθεστώς της χώρας στην οποία βρίσκονται. Πρέπει λοιπόν να εκριζώσουμε τις βαθύτατες αιτίε της τρομοκρατίας, να σταματήσουμε επίσης την χρηματοδότησή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεργαστούν ακόμα περισσότερο. Μπασίρ, ένα λεπτό. από το Πεσαβάρ στο Παρίσι και από τις Βρυξέλλες στη Λαχώρη. Εγώ πάντα καταδίκαζα την τρομοκρατία. Είναι ανεξήγητες και ασυγχώρητες ενέργειες βαρβαρότητας που δεν μπορεί να δικαιολογηθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό που έγινε στη Λαχώρη δεν θα πρέπει να είναι διαφορετικό. Πρέπει με ένα απλό μήνυμα να καταδικάσουμε τα εγκλήματα αυτά και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Όχι όροι, όχι προϋποθέσεις. Δυστυχώς κάποιοι ε, χρησιμοποιούν ε, αυτή την ευκαιρία για να δώσουν μαθήματα στο Πακιστάν για τα εσωτερικά του θέματα. Σκεφτείτε μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν στην Ευρώπη μια άλλη χώρα να μας έλεγε ότι λυπάμαι αλλά οι μεταναστευτικές σας πολιτικές και οι πολιτικές καταπολέμησης του, κοινού, του κοινωνικού αποκλεισμού οδήγησαν σε αυτό το οποίο έγινε. Μη με παρεξηγείτε. Ε, προφανώς θα πρέπει να γίνει συζήτηση για το Πακιστάν αλλά δεν είναι η σωστή στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ο κύριος Βόμποντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Καλωσορίζω το ψήφισμα διότι καταδικάζει αυτή τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση της οποίας τα θύματα ήταν σε μεγάλο βαθμό χριστιανοί αλλά και μουσουλμανοί. Είναι η κοινότητα που διώκεται περισσότερο, ε, κατατρέχεται περισσότερο με τον κόσμο και θα πρέπει να τους υπερασπιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος είναι ο στόχος με τα ψηφίσματα για τα κατεπήγοντα. Όχι για να καταγγέλουμε την κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάποιες χώρες, αλλά για να ε, φέρνουμε στην επιφάνεια τις απειλές που δέχονται συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Σημείο 9 του ψηφίσματος, η BB ε, ε, καταδικάστηκε σε θάνατο για βλασφημία και όχι για ε, τρομοκρατία και περιμένει στη φυλακή εδώ και 6 χρόνια την εκτέλεση της ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι εκκλήσεις δεν παραμένουν κενό γράμμα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καρυμή, ένα λεπτό. Μπορεί κανείς ε, να πηγαίνει στον ναό του ή στο τζαμί του ελεύθερα στο Πακιστάν. Αυτό δεν έχει ουδεμία σχέση με το Πακιστάν. οποιοδήποτε σκοτώθηκε ή ακροτηριάστηκε σε αυτές τις επιθέσεις είναι Πακιστανός. Αν είναι να τους διαχωρίζουμε σε κατηγορίες το ψήφισμά μας, προσβάλλουμε τη μνήμη τους. Κράτη και δρόντες που στηρίζουν τα τρομοκρατικά δίκτυα θα πρέπει να ξέρουν. Αποκαλύπτεστε. Θα συλληφθείτε και θα εκτεθείτε εντελώς οι τρομοκρατικές επιθέσεις είτε στη Λαχώρη, είτε στο Λονδίνο, είτε στις Βρυξέλλες ε, είναι επίθεση σε όλους μας και στεκόμαστε στο πλευρό τους για να τους αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βουλευτά. Τελείωσε λοιπόν αυτή, ε, αυτός ο καταλόγος Περνάμε στο Catch the Eye. Έχετε τον λόγο, συνάδελφε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τους προηγούμενους ομιλητές που καταδίκασαν όλη την τρομοκρατία. Είναι όμως απαραίτητο από την Ευρώπη να υπάρξει μια ξεκάθαρη προειδοποίηση ότι ναι μεν πρέπει να προασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά όχι μόνο στο χαρτί αλλά και στην πραγματικότητα. Πρέπει να το πούμε αυτό και στην πακιστανική κυβέρνηση. Περιμένουμε από πλευρά στι συγκεκριμένε ενέργειε για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καθημερινότητα τη ζωή στη χώρα αυτή. Αναφέρομαι στο θέμα αυτό όχι μόνο λόγω των καταστάσεων των θρησκευτικών διακρίσεων αλλά και εθνοτικών διακρίσεων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και να μην το ξεχνάει κανείς ότι έχουμε προβλήματα στο Βαλουχιστάν επί τη βάση πολλών πληροφοριών της Διεθνούς Αμνηστίας η Ευρώπη πρέπει να διευκρινίσει τα πράγματα, να δούμε τι είδους διακρίσεις υπάρχουν, όχι θρησκευτικέ μόνο, αλλά εθνοτικές. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι άνανδρες τρομοκρατικές επιθέσεις κατά χριστιανών την Κυριακή του Καθολικού Πάσχα στη Λαχώρη μας θυμίζουν ότι η Ισλαμιστική τρομοκρατία δεν χτυπάει μόνο την Ευρώπη οι επιθέσεις αυτές κόστισαν τη ζωή σε πάνω από 70 ανθρώπους δηλαδή περισσότερος από ό,τι στις τρομοκρατικές επιθέσεις στις βρυξέλλες. παρ' όλα αυτά δεν φάνηκε αυτό να ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ευρώπη. όταν η ευρωπαϊκή ένωση δεν καταφέρνει να διαχειριστεί τους εκτοπισμένους του εμφυλίου της συρίας που είναι μια χώρα 20 εκατομμυρίων καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε περίπτωση αποσταθεροποίησης του πακιστάν των 200 εκατομμυρίων κατοίκων το ενδεχόμενο γενικευμένης αποσταθεροποίησης σε μέση ανατολή και κεντρική ασία πρέπει να αποτραπεί πάση θυσία. για αρχή θα πρέπει να πάψουν οι στρατιωτικές επεμβάσεις των ξένων. επίσης θα πρέπει να πάψουν οι υπηρεσίες των δυτικών χωρών να παίζουν με τη φωτιά στηρίζοντας εδώ και εκεί οργανώσεις ισλαμιστών προς εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων στόχων. τέλος θα πρέπει να στηριχτούν όλες οι προσπάθειες που επιχειρούν έντιμα να υπερβούν το διαθρησκευτικό μίσος και τη ρητορία της πολιτισμικής σύγκρουσης. Ehm, ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. αυτό το οποίο συνέβη το πάσχα στο πακιστάν είναι κάτι το οποίο διέπραξε η ισλαμική τρομοκρατία αλλά να μην ξεχνάμε, να μην ντρεπόμαστε να πούμε ότι οι τρομοκράτες οι Ισλαμιστές σκοτώνουν τους χριστιανούς επειδή είναι χριστιανοί. Και τι κάνουμε εμείς, εμείς σαν ζόμπι κοιτάμε γύρω μας και δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Σκοτίστηκαν οι μεγάλοι Ευρωπαίοι πολιτικοί γιατί ποτέ δεν μπαίνουν στα μετρό, ποτέ δεν πηγαίνουν στις αίθουσες των αεροδρομίων να κάνουν ώρα έχουν τα δικά τους ιδιωτικά μέσα μεταφοράς. Οι απλοί πολίτες όμως φοβούνται για αυτά τα οποία συμβαίνουν και εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Εμείς αδιαφορούμε. Μπορούμε να σκοτώνουμε χριστιανούς ή Ισλαμιστές τρομοκράτες, θα πρέπει να τιμωρηθούν όμως και με την ποινή του θανάτου. Η Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στον συνάδελφο ότι σαν Ευρωπαία πολιτικός εγώ παίρνω το μετρό και εγώ κάνω ουρά στα αεροδρόμια όπως όλοι οι πολίτες. Όμως νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταδικάσει την τρομοκρατία η οποία ε, υπάρχει εις βάρος θρησκευτικών ομάδων στο Πακιστάν. Εμείς προσκαλούμε την κυβέρνηση του Πακιστάν να καταπολεμήσει αυτές τις βίαιες ομάδες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αναφέρθηκε η περίπτωση της Αϊσά Μπίμπι. Πρέπει να απελευθερωθεί η γυναίκα αυτή. Το ζητάμε εδώ και ε, πολλά χρόνια. Περιμένει τη θανατική της εκτέλεση και εμείς το καταδικάζουμε. Αυτό είναι μια γυναίκα που δεν έκανε τίποτα το λάθος. Απλά εξέφρασε ε, μια ελεύθε, με ελεύθερο τρόπο την πίστη της, το δικαίωμά της δηλαδή για την ελεύθερη πίστη και εξομολόγηση. Δυστυχώς όλα αυτά διώκονται ποινικά στο Πακιστάν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η θρησκευτική παράδοση εορτασμού, το Πάσχα, ε, με, ε, μετα, Τράπηκε σε τραγωδία. 73 πέθαναν, εκ των οποίων 13 παιδιά. Ε, ε, να άλλη μία απόδειξη για τις διαστάσεις αυτού του ανεξάρτητου μίσους κατά των ε, της χριστιανικής κοινότητας και δεν ενδιαφέρει τους Ισλαμιστές ότι οι θύματα ήταν και μουσουλμάνοι. 2% του πληθυσμού είναι χριστιανοί ε, στο Πακιστάν και αυξάνονται οι επιθέσεις εναντίον τους. Ε, στη Λαχώρη υπήρξε ήδη μια τρομοκρατική επίθεση με 17 θύματα. Κάνουμε ένα μικρό βήμα με το σημερινό ψήφισμα, όμως δεν έχει νόημα αν δεν έχουμε και δράση παρακολούθησης. Δεν υπάρχουν σύνορα για τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές, να ζητήσουμε από την Ισπανικαστική Σύγκριση επίσης την απελευθέρωση της Άσης Αμπίμπη. Ε, παρακαλώ. Ο κύριος Κέλλη. Νομίζω ότι οι επιθέσεις στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι αλλά και στο Πακιστάν δείχνουν, ε, έχουν αυτό το κοινό ότι δείχνουν τα πόσα υποφέρουν οι άνθρωποι ανά τον κόσμο και τι πρέπει να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε την ε, τρομοκρατία. Ε, υπάρχει αυτός ο ιδεολογικός πόλεμος κατά του εξτρεμισμού που έχει εξίσου μεγάλη σημασία όπως και η καταπολέμηση των τρομοκρατικών επιθέσεων. προσπαθούν οι κυβερνήσεις να θεσπίσουν μεταρρυθμίσεις κυρίω ε, κυρίως ε, για την κατάργηση των καταναγκαστικών γάμων και την προστασία ε, των ανθρώπων κατά της διακριτικής μεταχείρισης. Δεν φτάνουν όμως αυτά. Χρειαζόμαστε περισσότερα για να ασκήσουμε πίεση στις κυβερνήσεις αυτές, ούτως ώστε πέρα από τις μεταρρυθμίσεις ε, να υπάρχει και εφαρμογή των νέων διατάξεων, η υπερβολική διακριτική μεταχείριση κυρίως ε, κατά των γυναικών, κατά των ε, θρησκευτικών μειονοτήτων που προσιλητίζονται στο Ισλάμ λόγω των καταναγκαστικών γάμων και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι πέρα από το χέρι μας για να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Τελειώσαμε τώρα με τους ομιλητές και θα ακούσουμε την ε, κυρία Τάισεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Όπως και στο Πεσαβάρ, έτσι και στη Λαχώρη, η επίθεση την Κυριακή του Πάσχα στο στα παιδιά, στο μέλλον της χώρας η επίθεση της Λαχώρης είχε στόχο να σκοτώσει χριστιανούς, σκότωσε και πολλούς ε, μουσουλμάνους βεβαίως. Η επίθεση αυτή έρχεται μόλις δύο χρόνια μετά τους πουμαρτισμούς εκκλησιών πάλι στη Λαχώρη. Η συναδελφός μου, η Φεντερίκα Μοργερίνη, είπα πατή εκπρόσωπος, ε, εξέφρασε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και την στήριξή μας στο Πακιστάν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ζητάμε από το Πακιστάν να φέρει τους δράστες ε, και τους υποκινητές ε, της επίθεσης αυτής στην δικαιοσύνη. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για το αυξανόμενο επίπεδο θρησκευτικής βίας ε, και έλλειψης ανεκτικότητας στο Πακιστάν. Και Βεβαίω παρακολουθούμε τις δραστηριότητε. Ε, οι μειονότητες και οι θρησκευτικέ μειονότητες στη χώρα υποφέρουν δυσανάλογα και είναι συχνά στόχο των ακραίων. Ζητάμε από την κυβέρνηση να ενισχύσει τις προσπάθειες για να εξασφαλίσει την, την ε, σωματική ασφάλεια όλων των χωρικών και όλων των μειονοτήτων και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας απασχολούν πάντοτε στον τακτικό διάλογο με το Πακιστάν και καλούμε τις αρχές να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις δεδομένων αυτών των δύσκολων συνθήκων που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται για την άρση του μορατόριου μας προς την εκτέλεση της θανατικής ποινής και τον αριθμό των εκτελέσεων που έχουν λάβει χώρα και που φέρουν τώρα το Πακιστάν στην τρίτη καταθέση σειρά στις χώρες που εκτελούν τη θανατική ποινή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν καταδικάζει τη θανατική ποινή σε κάθε περίσταση και με επιμονή ζητεί την κατάργησε τη σε όλο τον κόσμο. Σε όλες τις επαφές της με το Πακιστάν η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υπογραμμίσει την σημασία της επανεισαγωγή του μορατόριου στι εκτελέσεις και τη στήριξη ελάχιστων προδιαγραφών. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει διάφορα έργα για την ενίσχυση τη ευαισθησία της πρόσβασης ε, στη δικαιοσύνη, της γνώσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ενίσχυση των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Πακιστάν. Η διμερής ε, συνεργασία για την ανάπτυξη 2014-2020 με 645 συνολικά εκατομμύρια ευρώ έχει στο επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα και την χρηστή διακυβέρνηση οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν ευρέ, ευρέως στη χώρα παρά τις κάποιες ε, προόδους υπάρχουν προόδοι για το θεσμικό πλαίσιο στο Πακιστάν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, παραδείγματι, έχει θεσπιστεί μια Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και επιπλέον, η κυβέρνηση πρόσφατα υιοθέτησε πρόγραμμα δράσης για τη βελτίωση της καταστάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν με διάφορα μέτρα ιδιαίτερα ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Δράση έχει επίσης αναλυφθεί για την αντιμετώπιση του ευρέως δεδομένου προβλήματος της ρητορικής μίσους και εισάγεται και σχετική νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης απευθύνει εκκλήσεις για μια συνολική δράση κατά της ε, τρομοκρατίας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, τις θεμελιώδεις αξίες και τις διεθνείς προδιαγραφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη της τρομοκρατίας και δι στους τομείς ε, αντιμετώπισης της ρωσοσπαστικοποίησης, ε, των επιστρατεύσεων, των στρατολογήσεων καλύτερα και τη πρόληψη τη τρομοκρατία γενικά. Πρέπει να υπογραμμίσω κυρίε και κύριοι πω η Ευρωπαϊκή Ένωση ήτο και παραμένει ε, στεναρός τη της ε, δημοκρατίας και των μεταρρυθμίσεων στο Πακιστάν. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λάβει